So, <clears throat> dear colleagues, dear guests. Συνάδελφοι προσκεκλημένοι, είμαστε πολύ λίγοι βουλευτές εδώ, αλλά ούτως ή άλλως πρέπει νομίζω να αρχίσουμε. Αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει μια αλλαγή, προσέξτε παρακαλώ. Δυστυχώς ο κύριος Ήβαν δεν μπορεί να έρθει σήμερα για το σχέδιό του για τις νέες τεχνολογίες και τις ανοιχτούς πόρους παιδείας, εκπαιδευτικούς πόρους. Αύριο το πρωί όμως θα έρθει. Προτείνω λοιπόν σήμερα να κάνουμε το 4, το 4 αύριο το πρωί ως πρώτο θέμα μετά τις ψηφοφορίες. Με αυτή την αλλαγή εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται. Εντάξει. Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2013. Τα έχετε στους φακέλους σας. Προτείνω συνήθως αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να θεωρηθούν εγκριθέντα. Τώρα για τη σημερινή διερμηνία έχουμε πολλή διερμηνία σήμερα αλλά δεν έχουμε τσεχικά και καμία βαλτική γλώσσα. αλλά ούτε τις χρειαζόμαστε. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, το 4 αναβάλλεται για αύριο και άρα περνάμε στο 5. Δημόσια ακρόαση, νέες τεχνολογίες και ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Σήμερα όπως μόλις σας είπα, έχουμε δημόσια ακρόαση με θέμα νέες τεχνολογίες και ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζει η Επιτροπή μας. Η ψηφιακή επανάσταση αφορά πλέον όλες τις πτυχές της ζωής μας, μεταξύ των οποίων και την παιδεία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν το κόστος της παιδείας και να προωθήσουν πιο ευέλικτους τρόπους μάθησης. Τελευταία, σημειώθηκε τεράστια αύξηση μαθημάτων και άλλων πόρων που διατίθενται από το Ιντερνετ είτε δωρεάν ως ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη είτε ως πληρωνόμενη πόρη. Αλλά η Ευρώπη δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα στο μέγιστο αυτές τις νέες τεχνολογίες ούτε αυξήθηκε πάρα πολύ σημαντικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του ίντερνετ. Η έκθεσή μας θα κάνει συστάσεις για το πώς θα μπορούσε η Ευρώπη να βελτιώσει αυτή την κατάσταση, να ανοίξει την παιδεία, να εφαρμόσει πιο καινοτόμες μορφές διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και περισσότερη χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε μια πρώτη ανακοίνωση της Κομισιόν, όπου καθορίστηκε ένα πρόγραμμα για τη χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας και των εκπαιδευτικών πόρων εκεί ταύτιζε αλλαγές σε τρεις τομείς. Καινοτομία στην παιδεία και στην εκπαίδευση, δεύτερον τη χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και τρίτον τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών πόρων και εγκαταστάσεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας. Πρώτα ο κύριος Κλάβδιος Ντόντι που είναι μέλος της συμβουλευτικής ομάδας της Κομισιόν για την ε, τεχνολογία της εκπαίδευσης. Δεύτερον, ο κύριος Βίλεμ Φαν Φάκελμπουργκ, που είναι συντονιστής της TU στο Delft, των ηλεκτρονικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο Delft. Και τρίτον, ο κύριος Χάουαρτ Μέγερ, που είναι διευθυντής και εκδότης στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες, τον καθένα για 10 ή 15 λεπτά, αλλά όχι περισσότερο, αλλιώς θα παρέμβω. Και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε να, αυτά που είπαν οι εμπειρογνώμονες για 40 λεπτά και ύστερα οι εμπειρογνώμονες θα απαντήσουν και τέλος θα λάβει το λόγο κάθε φορά θα το λόγο η Κομισιόν. Δίνω λοιπόν πρώτο το λόγο στον κύριο Ντόντι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα αξιότιμα μέλη. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα εδώ να σας μιλήσω στα πλαίσια της δημόσιας ακρόασης. Ο τίτλος είναι μία αναδιατύπωση ενό σημείου του σχεδίου έκθεσης, το 2 του Κοινοβουλίου, της έκθεσης του Κοινοβουλίου, που λέει ζητεί από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν οργανωτικό περιβάλλον στο οποίο τέτοιες καινοτομίε θα είναι ευπρόσδεκτες. Και έδωσα και εγώ τον τίτλο στην ομιλία μου τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι έτοιμα να ε, δεχθούν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και καινοτομίες στην τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας. Αυτή την εποχή όσοι έχουν αφιερώσει χρόνο στους πειραματισμούς, στην εκπαίδευση και την τεχνολογία χαίρονται που βλέπουν ότι υπάρχει ανανέωση της δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, στην ανοιχτή εκπαίδευση και στην τεχνολογία πληροφορίας επικοινωνίας. Η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικό βήμα προς τα μπρος και στηρίζει την τεχνολογία πληροφορίας εκπαίδευση και ανοιχτή εκπαίδευση. Είναι σημαντικό βήμα μπροστά, όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο έγγραφο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επειδή έχει στρατηγική αξία, αναφέρεται στον ευρύτερο στόχο της εκπαίδευσης, αναφέρεται στην ποιότητα. Δηλαδή, η ΑΕΠ, οι τύποι έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ποιότητα, να την αναβαθμίσουν, όχι εκπαίδευση στο ίδιο επίπεδο. Η συνολική εκπαίδευση και κατάρτιση αναβαθμίζονται. Αυτό έχει σημασία γιατί οι τεχνολογίες χρειάζονται στην κοινωνία μας και μπορούν να συμβάλλουν ε, στην καθημερινή ζωή μας, στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εκπαίδευση με παρόμοιο τρόπο. Αποτελεσματικότητα. Καμιά φορά ε, την υποτιμούμε, αλλά βέβαια η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε νέους τρόπους οργάνωσης ε, των οικονομικών της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τέλος, ε, ισότιμη πρόσβαση, κατάργηση αποκλεισμών, άνοιγμα της εκπαίδευσης που άρχισε μετά τα ανοιχτά πανεπιστήμια. Διαφέρει από τα άλλα κείμενα όπου επιμέναμε στις ε, δυνατότητες ε, των ΤΠΕ για την πρόσβαση ή την επιτάχυνση της απόκτησης ε, δεξιοτήτων αυτό είναι πιο ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τα μεγάλα ερωτήματα όμως είναι αυτά, αυτό το έγγραφο και τα σχετικά όπως το σχέδιο έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αρκετά για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν, το υπογραμμίζω αυτό το διατηρήσουν γιατί αυτό είναι ο αδύναμος κρίκος μάλλον, να διατηρήσει την ε, προσοχή εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε όλα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σχετικά με τη συστημική δυναμική των TPE να ε, αλλάξουν ποιοτικά τις αλλαγές θα υπάρξουν αντίκτυποι μόνο σε επιμέρους ε, τομείς του συστήματος της εκπαίδευσης. Η φιλοδοξίες ε, συνδέονται και με άλλα μέσα και μηχανισμούς που μπορούν να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν αλλαγές μέσα από τη χρήση των ε, ΑΕΠ, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων δηλαδή. Θα υπάρξουν δηλώσεις χωρίς όμως να συνοδεύονται από ε, μέσα πολιτικά. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιες θεμητές αμφιβολίες γιατί κατά το παρελθόν η προσοχή των πολιτικών στην χρήση των ε, ΤΠΕ χρησιμοποιούσε βραχείς κύκλους. Μετά από κάνα δυο κύκλους υπερβολών και προσέλκυση ενδιαφέροντος ε, μειωνόταν η προσοχή σε όλα αυτά και εστίαζαν σε άλλα προβλήματα που αφορούσαν εκπαίδευση, κατάρτιση, διαβίου, μάθηση κλπ και η συστημική θεώρηση του πώς οι τύποι ε μπορεί να ασχοληθούν με το θέμα της διακοπής της εκπαίδευσης ή της συμμετοχής των ενηλίκων σπουδαστών. Και οι σημαντικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την ε, αξιολόγηση της επιτυχίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος ε, δεν εξετάστηκαν. Μπορεί εκείνοι που εργάζονται στον τομέα να μην εξηγούν την κατάσταση πολύ καλά ή τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Μπορεί να παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρκετά, απο, αρκετές αποδείξεις των θετικών εξελίξεων. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία μεγάλης κλίμακας του τι κάνουμε είναι ότι δουλεύουμε εμβαλωματικά. Δηλαδή πιάνουμε ένα θέμα κάθε φορά και όχι δεν πιάνουμε ε, συνολικά το θέμα. Πολλές φορές ε, οι επενδύσεις στην τεχνολογία έγιναν γρήγορα, εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ε, άλλα πράγματα όμως, άλλοι παράγοντες και συνιστώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη. Οπότε κατά κάποια έννοια δεν ήταν δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό που λέω τη σωστή θερμοκρασία για να αρχίσει μια αλλαγή. Σε πολλές διαδικασίες χρειάζεται να φτάσουμε σε μια θερμοκρασία στη φυσική, στη χημεία, στις διαδικασίες εκεί. Και στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς χρειάζεται να φτάσουμε στη σωστή θερμοκρασία, η οποία ε, επιτυγχάνεται όταν έχουμε φύγει από τις υπερβολές και πριν κρυώσουν τα πράγματα. Ε, δηλαδή εκεί είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιτεθεί σωστή θερμοκρασία. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και η απαραίτητη μετατροπή όλων των θεσμικών παραγόντων, όλων που λαμβάνουν αποφάσεις σε επίπεδο κάθε σχολείου, κάθε πανεπιστημίου, κάθε κέντρου εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε εξηγήσει και σε οργανωτικό επίπεδο. Σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που προβάλλονται για να εξηγηθεί η μέτρια χρήση των ε, ΤΠΕ. Σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται πολύ, υπάρχουν, ε, υπάρχει προθυμία. Αλλά πόσες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να αξιοποιήσουμε πλήρως την τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσουμε. Ε, ε, επίσης η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη χρόνου, η ικανοτήτων ε, των εκπαιδευτικών, έλλειψη υποστήριξη από τους εμπλεκομένους. Καμιά φορά λένε οι δάσκαλοι, εμείς δουλεύουμε και πάμε να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Οι γονείς όμως έρχονται και λένε ότι θέλουν τα παιδιά τους να επικεντρωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, αυτό στο οποίο θα εξεταστούν στο τέλος της χρονιάς. Επίσης είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι, τα δίκτυα, οι, όλοι δηλαδή, οι δάσκαλοι, οι γονείς, εργοδότες, όλοι αυτοί να γνωρίζουν την κατάσταση και να συμμετέχουν στην διαδικασία για να συμβάλλουν και αυτοί στον επιτευχθεί αυτό που είπαμε η σωστή θερμοκρασία. Ο συνδυασμός τριών παραγόντων κατ' εμέ και πάω στα συμπεράσματα χρειάζεται ώστε να ε, δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα η πολιτική μας. Θέλουμε ε, πολιτικές που διευκολύνουν την καινοτομία. Τώρα έχουμε πολιτικές που μιλάνε για την, και, για την καινοτομία. Ε, φιλόδοξα προγράμματα. Στη θεωρία όμως. Αλλά μας λείπουν πολιτικές ως επιτοπλίστων που συμβάλλουν στις αλλαγές, από το πώς είναι φτιαγμένα τα νέα προγράμματα διδασκαλίας μέχρι ε, όπως ε, χτίζεται η εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση των ε, εκπαιδευτικών, πλαίσια για τη διασφάλιση ποιότητας, ένα κεντρικό θέμα στην έκθεση του Κοινοβουλίου, που πολύ σωστά το αναδεικνύεται και το λέει και η ανακοίνωση της Κομισιόν, είναι ότι χρησιμοποιούμε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θεωρεί τις ΤΠΕ ως μια ειδική αγορά αν θέλετε, ε, μια, ε, ε, έναν ειδικό τομέα που δεν καλύπτει όλη την εκπαίδευση. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν και ορισμένα κριτήρια που προστίθενται στα μοντέλα διασφάλισης ποιότητας, αλλά δεν υπάρχει μια πλήρης επανεξέταση της διασφάλισης ποιότητας στο φως του τι μορφή έχει η παιδεία στον αιώνα μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να ζητάμε από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να είναι έτοιμα να αλλάξουν όταν υπόκεινται σε περιορισμούς όπως τα παλιά προγράμματα διδασκαλίας κλπ. Ε, τα οποία εστιάζονται στις εξετάσεις. Η αξιολόγηση της μάθησης είναι πολύ ε, σημαντικό θέμα. Εκεί πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν μπορεί να περιοριζόμαστε σε εξετάσεις στο τέλος του έτους όπως τις έχουμε μέχρι τώρα, γιατί έτσι δεν μπορεί να προωθηθεί η εκπαίδευση μέσα από την αξιολόγηση. Ούτε θα χρησιμοποιηθεί πλήρως η τεχνολογία για να αναλύσει τη συμπεριφορά των ε, μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Ενώ ε, αυτό μπορεί να το κάνει η τεχνολογία. Αυτό λοιπόν είναι ένα. Ε, πολιτικές που θα διευκολύνουν τις καινοτομίες. Δεύτερον, ε, η ηγεσία που θα προσανατολίζεται στο, στην καινοτομία σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δηλαδή να είναι ε, ένα δίκτυο το οποίο θα επενδύει στο μετασχηματισμό σε επίπεδο πανεπιστημιακό Υπάρχει μια ευαισθησία στο θέμα αυτό, δηλαδή ξέρουν ότι ακόμα η τύπη δεν είναι κομμάτι της διαδικασίας της Μπολόνια, είναι πολύ περιθωριακός ακόμα ο ρόλος τους και αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Η τρίτη προϋπόθεση είναι η υποστήριξη στο δίκτυο συνεργασίας των καινοτόμων ε, εκπαιδευτικών. Ε, τη ηλεκτρονική αδελφοποίηση, για παράδειγμα, υπάρχει για τους δασκάλους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην εκπαίδευση και πρέπει με συστηματικό τρόπο να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς στη βάση. Με μαζικότητα αυτό είναι σημαντικό. Τονίζεται τους τελευταίους μήνες. Και τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μεγάλη ανάγκη να υποστηριχθεί η μικροκαινοτομία που προέρχεται από τη βάση. Σε αυτό το επίπεδο θα κινητοποιηθούν μεγάλοι αριθμοί εκπαιδευτικών. Τέλος, ε, η δυνατότητα υποστήριξης πρωτοβουλειών ευρωπαϊκών μεγάλης κλίμακας από τα υπάρχοντα προγράμματα και τα ταμεία. Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί αν υπάρξει σύγκληση ε, των διαδικασιών και της θερμοκρασίας που είπαμε, ε, για να γίνει αυτό χρειάζονται εμβληματικά έργα, μεγάλα έργα, μεγάλες προσπάθειες που ίσως είναι δύσκολο να ενταχθούν στην παρούσα δομή του ε, προγράμματος Έρασμους. Το έρασμος 2020 διαφέρει, νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ να γίνει η προσπάθεια της σύγκλησης ορατή. Ε, πιλωτικά προγράμματα, ε, μικρά προγράμματα για ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε πιο συστημικά και να συμπεριλάβουμε στρατηγικές ε, πρωτοβουλίες που θα φαίνονται όπως η αδελφοποίηση των σχολείων και έτσι θα γίνουν ένα σημείο αναφοράς μέσω και βράχη πρόθεσμα. Είναι σημαντικό πάντως ε, μέσα από αυτή τη στήριξη που εκφράζει η κοινότητα τώρα στη χρήση της ανοιχτής εκπαίδευσης και των τεχνολογιών πληροφορίας και ε, επικοινωνίας είναι ε, να μην ξεχάσουμε το θεμελιώδη ρόλο των εκπαιδευτικών. Αλλάζει ο ρόλος τους, αλλά παραμένει θεμελιώδης. Οι προσαρμοσμένες, ε, εξατομικευμένες δυνατότητες πρέπει να διατηρηθούν. Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνίσταται σε μεγάλο βαθμό στην προσωποποιημένη μάθηση. Ό,τι είναι μαζικό θα πρέπει να μπορεί και να προσωποποιείται, να εξατομικεύεται. Τέλος, για τη χρήση των ΤΠΕ στον τομέα της ε, θεσμοθέτησης της ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε τώρα τα μαζικά αυτά διαδικτυακά μαθήματα που οδηγούν σε μοντέλα. Ένα, ένα πανεπιστήμιο με βάση αυτό το μοντέλο διανέμει τη γνώση, ως των αμερικανικά πανεπιστήμια είναι αυτά που διαχέουν γνώση, αλλά και τα ευρωπαϊκά αρχίζουν τώρα να μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι και μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω από το να αναπαράγουν αυτά τα μοντέλα τα μαζικά, των μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων. Και έχουμε και τη διαδικασία της Μπολόνια. Μπορεί και εκεί να υπάρχει σε αυτά τα πλαίσια συνεργασία και συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων. Μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτή τη συνεργασία ε, που στηρίζεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία για να έχουμε την εικονική ε, κινητικότητα ως, ένα, ε, ως μια προσέγγιση ευρωπαϊκή που θα είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο στο διανεμητικό μοντέλο της εκπαίδευσης. Αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε τούτη την ώρα και εφιστώ την προσοχή του ακροατηρίου μου εδώ ε, στις δυνατότητες που μπορεί να υπάρξουν. Θέλουμε λοιπόν κρίσιμη και υπεύθυνη και κριτική και υπεύθυνη ε, προσέγγιση να ξέρουμε ότι η ΑΕΠ και τα ΤΠΕ e δεν θα μειώσουν σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης για τις κυβερνήσεις, αλλά μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης για τους πολίτες. Το στοιχείο της πρόσβασης είναι μια μεγάλη αξία που σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί εμβληματική για το, την κίνηση αυτή, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πέσει η ποιότητα και η σημασία όλων αυτών. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι όλα αυτά και η χρήση της τεχνολογίας πέρα από τη διασφάλιση της πρόσβασης ε, και κάποια οικονομικά στοιχεία διατηρούν την ποιότητα και τη σημασία της εκπαίδευσης σε υψηλό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόντι. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Βαν Βάλκεμπερ, παρακαλώ. το μικρόφωνο. Ωραία. Ο τίτλος της παρουσίασή μου είναι λίγο πιο προκλητικός. Λέμε ότι το μέλλον της εκπαίδευση είναι διαδικτυακό. Δεν θα είναι απλώς και μόνο διαδικτυακό, αλλά το λέω έτσι, με την τιμή των όπλων. Είμαι υπεύθυνο στο Πανεπιστήμιο για την ανοιχτή και διαδικτυακή εκπαίδευση και επίσης συμμετέχω και στο Consortium Open Courseware και είμαι και Project Manager στο Open Courseware Europe. Αν δούμε λίγο το μέλλον, ο αριθμός των ε, φοιτητών ε, αναμένεται να τετραπλασιαστεί ε, στα 400 εκατομμύρια το 2030 σε σχέση με τα 100 που είχαμε το 2000. Αυτό βέβαια Ε, θα δημιουργήσει και προβλήματα διότι και οι φοιτητέ αναμένουν διαφορετικά πράγματα πλέον από το Πανεπιστήμιο. Καθημερινά χρησιμοποιούν το Facebook, το WhatsApp, το Google, το Twitter και όλες αυτές τις ε, διαδικτυακές πλατφόρμες και εμεί διδάσκουμε ακόμα στο μαυροπίνακα. Ε, έχετε εδώ μια φωτογραφία από το πανεπιστήμιό μου και νομίζω ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια αυτό είναι ο κατεξοχήν τρόπο διδασκαλία και αυτό φυσικά θα πρέπει να αλλάξει. Τα τελευταία δύο χρόνια ε, είδαμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα λεγόμενα MOOCs. Έχετε εδώ κάποιες ε, ε, ετικέτες και εγώ είμαι πολύ θετικός σε όλα αυτά, διότι θεωρώ ότι ο κόσμος αρχίζει πλέον να προσέχει τι ακριβώς συμβαίνει. Τι είναι όμως ένα MOOC. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί, οι οποίοι ε, ε, κυκλοφορούν για το MOOC και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε οποιονδήποτε όρο Οποιοδήποτε μάθημα γίνεται πλέον διαδικτυακά αποκαλείται MOOC, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για διαδικτυακή εκπαίδευση και όχι απλώς και μόνο ένα MOOC. Είπε ήδη ο προλαλής σας ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα λεγόμενα MOOCs και έχουμε πλέον πάνω από χίλια MOOCs διαθέσιμα διαδικτυακά, τα περισσότερα από αυτά από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, διότι εκεί υπάρχουν και οι μεγαλύτερες πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούνται και υπάρχουν και ευρωπαϊκέ πλατφόρμες, οι οποίε όμω είναι πολύ μικρέ. Υπάρχει το Future Learn στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα αντίστοιχο στη Γερμανία και το γαλλικό Νούμερικ από τα γαλλικά πανεπιστήμια. Όλα αυτά όμω σε πολύ μικρή κλίμακα προ το παρόν. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε μόνο τεχνικής φύσεως MOOC ε, όπω για παράδειγμα στη μηχανική, ενώ πλέον διατίθονται πάσης φύσεως μαθήματα μέσω MOOC. Τα MOOC Uh, Δεν είναι το παν βέβαια. Είναι ενδιαφέροντα διότι προσελκύουν πολύ το ενδιαφέρον των ε, ε, φοιτητών και όλοι στα πανεπιστήμια αναφέρονται στα MOOC και αυτό ίσως είναι ένας καλός τρόπος να διαδοθούν αλλά θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και πολύ περισσότερα πράγματα και αυτή είναι η διαδικτυακή επέδευση η οποία εδώ και 10 χρόνια κερδίζει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Έχω κάποια στοιχεία εδώ από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Το 2003 ήταν 11%, ενώ το 2011 έχουμε φτάσει ήδη στο 23% της διαδικτυακής διδασκαλίας. Φοιτητέ, δηλαδή που παρακολουθούν διαδικτυακά κάποιο μάθημα. Δεν έχω δει τα πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι έχει ανέβει κι άλλο το ποσοστό. Δεν γνωρίζω και τα στοιχεία στην Ευρώπη, μπορεί να τα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια, αλλά θεωρώ ότι υστερούμε σε αυτές τις εξελίξεις. Και θα πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε σε αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα εξαφαλιστεί. Τα MOOC δεν είναι μόδα που θα φύγει. Η διαδικτυακή εκπαίδευση εν γέννη είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα μείνει. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις ε, σχετικές εξελίξεις. Υπάρχει διαδικτυακή εκπαίδευση, υπάρχει τα MOOC, υπάρχουν ε, ναι. ανοιχτοί πόροι ε, παιδείας και υπάρχουν και προγράμματα τα οποία κινούνται διαδικτυακά. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Και η ορολογία είναι ανάμεικτη. Στο δικό μου το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι κυρίως πανεπιστήμιο ε, μηχανικής έχουμε ένα σλόγγαν, εκπαιδεύουμε τον κόσμο και βελτιώνουμε την ποιότητα της παιδείας. Αυτό ε, γίνεται εδώ και κάποια χρόνια και δεν θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για την έρευνα και για την ε, πληροφορική και την επικοινωνία, το ICT δηλαδή, να είμαστε ανοιχτοί σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αν δείτε λίγο το ε, πώς είναι κατανεμημένη η εκπαίδευση, περισσότερο έχουμε εκπαίδευση επιτόπου στο Πανεπιστήμιο, έχουμε 95% των φοιτητών οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά ε, και μεταπτυχιακά και έχουμε και διδακτορικούς φοιτητές ε, οι οποίοι όλοι βρίσκονται επιτόπου στο χώρο του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία ε, είναι και διαδικτυακά. Από το 2007 έχουμε 125 μαθήματα τα οποία διατίθεται διαδικτυακά, αλλά έχουμε και πάρα πολλέ ε, διαλέξει ε, οι οποίε διατίθεται στο διαδίκτυο. Υπάρχει και υλικό λοιπόν. Πέρσι ξεκινήσαμε με τα MOOC, είχαμε δύο MOOC, ένα για την μηχανική και ένα δεύτερο για την επεξεργασία των ιδέτων. Είχαμε περίπου 20.000 εγγραφές και δόθηκαν και 4.000 ε, πιστοποιητικά ε, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης αυτού του κύκλου μαθηματών και πλέον έχουμε ξεκινήσει και εξ αποστάσεως ε, προγράμματα από δύο σχολές του Πανεπιστημίου και ολοκληρώθηκαν 11 κύκλοι μαθημάτων. 50 φοιτητέ ενδιαφέρθηκαν για το θέμα αυτό και 30 εξ αυτών είναι ούτω ή άλλω φοιτητέ που προτιμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το μάθημα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται σε μία τάξη, αλλά προτιμούν να το κάνουν διαδικτυακά. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι όταν ξεκινάει κάποιο ένα εξ πρόγραμμα, δεν το κάνει για μια νέα ομάδα φοιτητών, αλλά και για του ήδη υπάρχοντε φοιτητέ, διότι το περιμένουν ότι θα υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία θα προσφέρονται από το διαδίκτυο. Ε, όλα αυτά προσφέρουν φυσικά μεταπτυχιακό τίτλο και υπάρχει πλήρης πιστοποίηση, επομένως αναγνωρίζονται. Αν δούμε τις πρόσφατες εξελίξεις και τις ε, ε, συγκρίνουμε με τις εξελίξεις, μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο με τις μεταφορές. Ξεκινήσαμε με την άμαξα, μετά είχαμε ένα κινητήρα, ο οποίος αφαίρεσε το άλογο, αλλά η ιδέα έμεινε ίδια και ε, η μεγάλη αλλαγή ήρθε με τα Ford, τα οποία ε, μπήκαν και σε μαζική παραγωγή και είχαμε ε, αυτοκίνητα, άρχισαν να παράγονται νέα μοντέλα, νέα δίκτυα και νέος τρόπος ζωής. Άρχισε πλέον ο κόσμος να μένει πιο μακριά από τη δουλειά του γιατί είχε την πελτέλεια να το κάνει. Και αν δούμε το μέλλον της παιδείας, ε, μπορούμε να το συγκρίνουμε αντίστοιχα με το πώς θα αλλάξει ο τρόπος ζωής στα πανεπιστήμια. Ε, τα πρώτα αυτοκίνητα είναι μια διάλεξη στην τάξη και η οποία απλώς μαγνητοσκοπείται και μετά προσφέρεται μέσω βίντεο στο διαδίκτυο. Τα MOOC για μας είναι τα πρώτα T-Ford αυτοκίνητα. στην πρώτη φάση των T4 είχαμε διάφορες εκδοχές και βλέπουμε και πολλές αλλαγές να γίνονται στα MOOC. Ε, αυτό θα δημιουργήσει νέα δίκτυα και το είδαμε ήδη αυτό με το Coursera και δημιουργούνται και νέες συμπράξεις που δημιουργούν δίκτυα νέων πανεπιστημίων που συνεργάζονται, ανταλλάζουν μαθήματα, χρησιμοποιεί ένα στα τα μαθήματα του άλλου και αυτό φυσικά θα συνεχιστεί. Και θα δούμε και νέα μοντέλα. Κάθε πανεπιστήμιο θα προσαρμόσει τα MOOC ε, με βάση συγκεκριμένα μαθήματα ή με συγκεκριμένο τρόπο. Κάποια πανεπιστήμια θα γίνουν ε, ε, οι δήμονες σε κάποια μαθήματα και θα δούμε και άλλες αλλαγές και θα αλλάξει και η ζωή μας. Θα υπάρχει πολύ περισσότερη διάδραση και θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και από πλευράς διαβίου μάθησης. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθεί κάποιος μαθήματα στο πανεπιστήμιο επειδή μπορεί να τα παρακολουθεί μέσω διαδικτύου και μπορεί φυσικά να ε, κάνει διάφορα πράγματα ταυτόχρονα. Ε, για το δικό μου το πανεπιστήμιο, τα επόμενα βήματα είναι ότι θα επεκτείνουμε και θα ξεκινήσουμε ένα διαδικτυακό πορτφόλιο. Θα προτείνουμε δηλαδή κάποια μαθήματα στα επόμενα δύο χρόνια θα αλλάξουν τα περισσότερα από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα και θα είναι είτε διαδικτυακά είτε μεικτά προγράμματα. Και επειδή ακριβώς επικεντρωνόμαστε και σε ε, αλλοδαπούς φοιτητές, όχι μόνο φοιτητές από την Ευρώπη αλλά από, και από όλο τον κόσμο, για παράδειγμα, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη διαχείριση των υδάτων έχουμε φοιτητέ από την Ινδονησία και την Αφρική και τους ενδιαφέρει το πρόγραμμα αυτό γιατί εμείς είμαστε προγνώμονες σε αυτό. Ξεκινάει και το DALF Extension School που είναι ε, ένα μοντέλο που θα έχει ε, διαδικτυακές ε, δραστηριότητες και το έχουμε αποκαλέσει έτσι για να θυμίζει το Harvard Extension School που είναι πολύ επιτυχημένο σε αυτή τη διαδικασία. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς αλλάζουν όλα αυτά. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και ένα κέντρο έρευνας και κοινοτομίας για την διαδικτυακή εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία, αλλά προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να το βελτιώσουμε. Τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια ε, δήλωση του Τόμας Φρίντμαν, ο οποίος λέει ότι όταν καταλα... αρχίζει να καταλαβαίνει ο καθένας τι συμβαίνει, τότε έχει τελειώσει μετριότητα. Και αν όλα τα πανεπιστήμια αρχίζουν να προσφέρουν τα καλύτερα του μαθήματα διαδικτυακά, γιατί να επιλέγουν οι φοιτητέ να έρθουν στο δικό σα το πανεπιστήμιο και γιατί να μην τα παρακολουθήσουν στο διαδίκτυο σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μέιτορ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι για την παρουσία μου. και για το ότι μου αφήσατε λίγο περισσότερο χρόνο οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες δεν θα τον χρειαστώ όλων. και θα συνεχίσω στα γερημανικά. Έχουμε λίγο χρόνο και σήμερα μιλάμε για μια εκτενέστατη πρωτοβουλία. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα. Και υπάρχουν ορισμένες πτυχές που δεν αναφέρθηκαν από τους δύο προηγούμενους ομιλητές. Αναφέρομαι στο σχολείο, ε, ψηφιακά σχολεία με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ψηφιοποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης, συμπερίληψη των επαγγελματιών στην ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων σε όλη αυτή τη διαδικασία της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος η πρωτοβουλία ανοίγματο της εκπαίδευσης εστιάζει πολύ στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ΑΕΠ, και επίση υπάρχουν και άλλε συνιστώσει που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Καταρχήν είναι σημαντικό να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει, την πρωτοβουλία πρέπει να την καλωσορίσουμε ιδιαίτερω και ελπίζω να υπερψηφιστεί από εσά. Ο κύριος Ντόντι ανέφερε ήδη ότι είχαμε σαφή υστέρηση απέναντι σε άλλες υπήρους και χώρες. Εμείς εδώ στην Ευρώπη, εις ό,τι αφορά τη χρήση ψηφιακών μέσων, ψηφιακών εξοπλισμών, ψηφιακών περιεχομένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό αναφέρεται στα έγγραφα και στις εκθέσεις ε, πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να αναλάβουμε δράση κατεπιγόντος, όχι για να μπούμε στο προσκήνιο των εξελίξεων, αλλά να καλύψουμε το χαμένο έδαφος απέναντι σε άλλες υπήρους και χώρες. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πολλά σημεία στην ανάλυση μας βρίσκουν σύμφωνος. Σε ορισμένα σημεία τα αίτια για τη σημερινή κατάσταση όμως δεν εξετάζονται στο απαραίτητο βάθος και έτσι μπορεί η σειρά μέτρων να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο για να επιτύχουμε συνολικά το στόχο του ανοίγματος της εκπαίδευσης πρέπει σαφώς να συμμετέχουν και να κινητοποιηθούν όλοι οι συμμετέχοντες ε, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να συνδεθούν οι σχολικές αίθουσες στο δίκτυο. Ε, θα πρέπει να οι στόχοι μάθησης να λαμβάνονται υπόψη γιατί είναι σημαντικοί για μία προσέγγιση ολοκληρωμένη. Όπως είπε ο κύριος Ντόντι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα μεμονωμένα περιορισμένη εμβέλεια προγράμματα, ούτω ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις που προανέφερα. Ε... Υπάρχουν ε, πολλοί ε, άξιοι εκπαιδευτικοί που έκαναν ε, ανάλυση των συστημάτων και θέλω να τους ε, συγχαρώ γιατί έλειπε μια εξέταση του συστήματος ε, εκπαίδευσης συνολικά στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στα ψηφιακά περιεχόμενα, θα πρέπει να μπορούν να τα επεξεργάζονται πιο εύκολα έτσι χρησιμοποιούνται με λογικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα σήμερα και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα ψηφιακά μηχανήματα, τα devices, οι συσκευές, είτε είναι tablets, οι mobile phones, οι smartphones, δεν έχουν και μεγάλη αξία αν δεν προβάλλουν περιεχόμενα. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι λοιπόν τα περιεχόμενα σε κεντρική θέση το άνοιγμα της εκπαίδευσης δεν πρέπει λοιπόν να στοχεύει μόνο στους ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη μόνο σε περιορισμένο βαθμό άλλες διαστάσεις. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα σχολεία, γιατί εκεί χάνουμε πολύ παραγωγικό δυναμικό. Οι ΑΕΠ δεν αποτελούν πανάκια απέναντι στις ε, ελλείψεις ε, που υπάρχουν ή ε, στις αδυναμίες που υπάρχουν στην αγορά. Στα σχολεία για 12-13 χρόνια συγκεντρώνονται όλοι οι μαθητές, ο μαθητικός πληθυσμός και οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι είναι σημαντικό ε, να υπάρχει συστηματοποιημένη μάθηση. Αυτά τα περιεχόμενα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Επίσης έχουμε ε, εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης που έχουν ε, πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά την προετοιμασία του μαθήματος. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν δεν έχουν χρόνο για να καταρτίζουν ε, το νέο αυτό υλικό, ιδιαίτερα σε επίπεδο τέτοιο που να μπορούν να το χρησιμοποιούν αυτό το υλικό και άλλοι εκπαιδευτικοί πολλοί επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο μέσα από ζητήματα όπως κατάργηση αποκλεισμών, ε, εξατομίκευση και το γεγονός ότι όλο και περισσότερο τώρα οι εκπαιδευτικοί ε, μεταφέρουν το μάθημά τους ε, στο ψηφιακό σύστημα. Ως επιτοπλίστων λοιπόν ε, οι προσπάθειες ε, περιορίζονται στο μάθημα που θα πρέπει ε, να διδάξουν μια συγκεκριμένη μέρα. Δεν έχουν μια συνολική προσέγγιση. Είπαμε λοιπόν ότι οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι δεν μπορούν να ε, αναπτυχθούν όπως πρέπει από τους εκπαιδευτικούς γιατί δεν έχουν χρόνο. Σε, ε, στη, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επειδή όμως υπάρχουν ποιοτικέ ελλείψεις ε, στο, εις δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το σύστημα δεν μπορεί να ε, εξελιχθεί όπως πρέπει. Ποιος θα ενημερώνει του ΑΕΠ, ποιος θα συμβάλλει ε, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής χρηματοδότησή τους. Πολλές φορές ε, περιοριζόμαστε σε projects τα οποία έχουν αρχή και τέλος και ξέρουμε από την πείρα μας με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μόλις τελειώσει η χρηματοδότηση ενός ε, έργου, ενός project, αυτό δεν χρησιμοποιείται πια, δεν το αξιοποιούν. Ε, είναι λοιπόν ε, ε, θέμα και γλωσσικό και πολιτισμικό ούτως ώστε να υπάρχουν δυνατότητες συνολικής αξιοποίησης αυτών των προγραμμάτων μην ξεχνάμε επίσης και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορούμε λοιπόν μόνο με τους ΑΕΠ να ε, διασφαλίσουμε αποτελεσματική και σύγχρονη λειτουργία των σχολείων. Ούτε θα επιτύχουμε την απαραίτητη κρίσιμη μάζα μαθησιακών εκπαιδευτικών περιεχομένων σε, με ψηφιακή, σε ψηφιακή μορφή. Η σύστασή μου είναι να στα πλαίσια της ε, πρωτοβουλίας άνοιγμα της εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τους ΑΕΠ, αλλά να ασχοληθούμε κυρίως με θέματα έρευνας και ανάπτυξης και να έχουμε συγκεκριμένους ΑΕΠ για τα σχολεία. Πολύ σημαντικό και χρήσιμο είναι να χρησιμοποιήσουμε και τους επαγγελματίες φορείς που προσφέρουν περιεχόμενα να ε, φροντίσουμε ούτως ώστε να συμμετέχουν άμεσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες ε, στα πλαίσια αυτών των πρωτοβουλειών. Έτσι εκπλήσει λίγο, αν δούμε με κριτικό ε, βλέμμα του ΣΑΕΠ, ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της ανάπτυξης και προετοιμασίας ε, περιορίζονται στις ακρογάσεις αλλά μετά όταν καταρτίζονται τα μοντέλα για την πρωτοβουλία δεν συμμετέχουν πια. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Εξίσου λυπηρό είναι το γεγονός ότι οι επαγγελματίες δημιουργοί συγγραφείς που υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες στην Ευρώπη που μέχρι τώρα έχουν αναπτύξει μαθησιακά μέσα για τα σχολεία ούτε αυτοί λαμβάνονται υπόψη. Καθόλου. Έχουμε καμιά φορά την εντύπωση ότι το υπάρχον μοντέλο μπορεί να είναι ελκυστικό για τον κλάδο ε, της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας, αλλά φαίνεται να συνιστά μια απειλή για την ε, βιομηχανία των μέσων, μέσων γενικότερα. Ε, δηλαδή η τεχνογνωσία, η αποτελεσματικότητα που υπάρχει ε, σε αυτούς τους τομείς ε, δεν λαμβάνεται υπόψη. Πολλές φορές ε, οι εμπειρίες περιορίζονται στα έντυπα μέσα και δύσκολα δημιουργείται η τεχνογνωσία για ψηφιακά προϊόντα και ψηφιακά μέσα. Η ανάπτυξη είναι αργή Ίσως γιατί δεν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο σχολείων, ούτως ώστε από τα έντυπα μέσα να περάσουν στα ψηφιακά. Οι εκπαιδευτικοί ε, δεν ε, παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη των ψηφιακών μέσων ή ε, δεν έχουν συμμετάσχει σε μέτρα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στα ψηφιακά μέσα. Ε, τα σχολεία επίσης δεν είναι αρκετά εξοπλισμένα και συνδεδεμένα στο διαδίκτυο ε, ή τουλάχιστον οι ταχύτητες των δεδομένων δεν είναι οι επαρκείς και έτσι δεν υπάρχουν επαρκή μέσα για εξοπλισμό σε ψηφιακά μέσα και περιεχόμενα ούτως ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή. Αυτό είναι ένα βασικό εμπόδιο και δεν εκπλήσει ότι τώρα η εκδοτική, οίκοι ε, δεν ε, δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη αυτών των περιεχομένων. Θέλουμε τώρα μια πρωτοβουλία που θα τα λαμβάνει υπόψη όλα αυτά. Επίσης, ε, στα πλαίσια των ΑΕΠ υπάρχει και ένα άλλο κεντρικό θέμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη δηλαδή. Πρόκειται για την προβληματική των λειτουργικών και βιώσιμων μοντέλων, δηλαδή πώς χρηματοδοτούνται οι ΑΕΠ μέχρι τώρα. Ε, είτε θα υπάρχει άμεση χρηματοδότηση δημόσια, εδώ υπάρχει και η Wikipedia ή η Kern Academy στις ΕΠΑ, υπάρχουν πολλοί σπόνσορες, και υπάρχουν και άπαξ προγράμματα χρηματοδοτούμενα τα οποία μπορεί να χρηματοδοτήσουν επιμέρους ε, συγγραφείς ή δημιουργοί. Εδώ υπάρχει ένα εναλλακτικό μοντέλο που θέλω να το παρουσιάσω σύντομα. Σημαντικό είναι καταρχήν να έχουμε τις απαραίτητες ε, προϋποθέσεις πλαίσιο, συνδεσιμότητα, ε, κομπιούτερ για κάθε μαθητή σε μια τάξη, ε, η σύγχρονη υποδομή, servers και όλα τα παρεπόμενα. Δεν σημαίνει ότι αν έχει ένα τάμπλετ στα χέρια του μαθητής θα έχει πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα και περιεχόμενα. Πρέπει επίσης να έχουμε και ε, εναλλακτικές ε, δυνατότητες. Αυτό είναι μια υπόθεση που στοιχίζει. Ο κύριος ε, ε, Φαν Φάλκενμπουργκ μας παρουσίασε πώς λειτουργεί το σύστημα στο πανεπιστήμιό τους. Στα σχολεία βέβαια δεν έχουμε φτάσει εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, να υπάρχει δικτύωση σε όλη την επικράτεια κάθε χώρα, στο σχολείο και πρέπει να κάνουμε διδακτική και παιδαγωγική έρευνα πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Όλοι οι παραγωγοί περιεχομένων πρέπει να συμμετέχουν, δηλαδή και ε, εκδοτικοί οίκοι και ε, φορείς που προσφέρουν πόρους, ε, περιεχόμενα, όλοι όσοι συμμετέχουν στην διαδικασία της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχουν. Υπάρχει ένα, μια πρόταση μοντέλου, δηλαδή ένα εθνικό εκπαιδευτικό δίκτυο το οποίο θα στηρίζεται ε, από όλους τους φορείς που προσφέρουν περιεχόμενα και τεχνολογίες και η λειτουργία του θα πρέπει να είναι να καλύπτει ε, ελλείψεις ε, στου σερβερ, στον κορμό, και, να κάνει εναρμόνιση περιεχομένων κλπ. Θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με τρόπο ανταπαδοτικό αλλά χωρίς κέρδος από, τις χρήστες, από τους χρήστες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους, ε, τις κοινότητες. Ε, αυτό το μέσον που θα είναι εναρμονισμένο θα το χρησιμοποιούν πολλοί φορείς, θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα ε, υπάρχει ε, μια δικτυακή πύλη. Έτσι θα κινούμεθα στα νομοθετικά πλαίσια που υπάρχουν και θα αποφεύγουμε στερευλώσεις του ανταγωνισμού. Θα υπάρχει μια ποιότητα ε, αξιολογημένη, ε, καταξιωμένη και θα εξασφαλίσουμε την ποιότητα μέσα από την συμμετοχή εκδοτικών οίκων και άλλων φορέων που προσφέρουν τέτοια περιεχόμενα. Θα διασφαλίζουμε έτσι υψηλή ποιότητα και θα ε, υπάρχει ανταγωνισμός για τους καλύτερους ΟΕΠ, ΑΕΠ. Ε, μια τέτοια λύση κατασκευάζομαι, είναι στα πρώτα της βήματα στη Γερμανία. Ε, επίσης ε, τα ψηφιακά περιεχόμενα μπορούν να ε, χωρίζονται σε ενότητες ε, ανάλογα με τις ανάγκες πολύ πιο εύκολα από ότι τα βιβλία. Θα μπορούμε έτσι να συνεργαζόμεθα πολύ περισσότερο με εκπαιδευτικούς φορείς άλλων χωρών. Αυτό δεν γίνεται εύκολο, εύκολα με βάση τα βιβλία. Και επίσης θα υπάρχει μέσα από το υγεία ανταγωνισμό ε, θα υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες ε, αξιοποίησης αυτού του μοντέλου. Ένα τέτοιο, παρακαλώ να ολοκληρώσετε, παρεμβαίνει και λέει η πρόεδρος. Ε, το φτιάχνουμε στη Γερμανία και συνεργαζόμεθα και με φορείς που προσφέρουν τέτοια περιεχόμενα. Τέλος, δείτε και την προοπτική της ε, σημειωτικής αναζήτησης ε, με το πρόγραμμα ανοίγματος της εκπαίδευσης ε, φτιάχνουμε και δικτυακές πύλες θα υπάρχουν σύντομα διαδικασίες για την σημαντική σημειωτική αναζήτηση, ούτως ώστε αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να προσφέρουμε παράλληλα περιεχόμενα, όταν υπάρχει αναζήτηση από κάποιον ενός περιεχομένου, ε, τα οποία θα είναι υποποηθητικά. Και τελευταία παρατήρηση. Ε, στηρίξτε μια κοινή δράση για την ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Εμείς θα συμμετάσχουμε όσο μπορούμε με την εμπειρία μας ε, και νομίζω ότι εδώ μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων των ε, εκδοτικών οίκων και των μέσων. Εμείς προσπαθούμε να συνεργαστούμε όχι μόνο στη Γερμανία με τους φορείς αυτούς, αλλά πανευρωπαϊκά και η πρωτοβουλία ανοίγματο της εκπαίδευσης παρέχει για μια τέτοια συνεργασία το ιδεώδες πλαίσιο. Ευχαριστώ οι συνάδελφοι τώρα θα μπορέσουν να παρέμβουν. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω εγώ δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση προς τον κύριο Βάλκενμπουργκ, διότι αναφερθήκατε σε μία τάση η οποία επικρατεί ε, το γεγονός δηλαδή ότι όλο και περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν πλέον ε, μαθήματα διαδικτυακά. Τι θα σημαίνει αυτό για τα πανεπιστήμια στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι κάποια τα οποία ε, δεν ε, είναι διατεθειμένα να προσφέρουν τέτοια μαθήματα θα εξαφανιστούν και τι γίνεται σε, από άποψη ανταγωνισμού μεταξύ των πανεπιστημίων που προσφέρουν τα καλύτερά τους μαθήματα διαδικτυακά και ποια όχι. Θα ήθελα λίγο περισσότερα από αυτού και εδώ θα κάνω την ερώτηση στα γερμανικά. Μας είπατε κύριε Μέλχερ ότι υπάρχουν και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα δημιουργού κλπ. που πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Έχετε λύσεις να προσφέρετε εδώ για το πώς θα λυθεί άπαξ και διαπαντός το πρόβλημα αυτό. Yes, Mr. for uh, question. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, ο κύριος Φάλκενμπουργκ. Εξετάζοντας ένα παραδοσιακό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη, ή τουλάχιστον στις κάτω χώρες, το 70% των μαθητών, των φοιτητών, ε, κατάγονται από την περιοχή στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο. Και υπ' αυτή την έννοια πολλά από τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν φυσικά να υφίστανται, αλλά δεν θα έχουν τους καλύτερους τους φοιτητές, διότι θα επιλέγουν οι φοιτητές να συμμετέχουν διαδικτυακά στο καλύτερο πανεπιστήμιο που μπορούν. You will get an, uh, I think a division between uh, regional universities and και από εκεί και πέρα τη σχέση μεταξύ των παραδοσιακών πανεπιστημίων και των ε, καλύτερων πανεπιστημίων, νομίζω ότι εκεί θα υπάρχει μια διάκριση. Η επόμενη σας ερώτηση... για τα ε, πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εκδοτών και το κατά πόσον μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου την εμπορική ε, αλλά και την τεχνική σκοπιά αυτών των ερωτημάτων σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο να αλλάξει η νομοθετική κατάσταση από αυτού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο αντίτιμο για όλους όσου προσφέρουν περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με ψηφιακή μορφή. Εάν επιληθεί αυτό το πρόβλημα, τότε ίσως μπορεί να επιληθούν και τα ε, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει πρώτα λοιπόν να λυθεί το θέμα του οικονομικού αντιτίμου και να υπάρχει κατάλληλη πληρωμή για τους εκδότες, για τους ε, ε, όσους ασχολούνται με τις τεχνικές λύσεις και από εκεί και πέρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να λυθούν και τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων. Βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία και χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε πιο κατάλληλες λύσεις για την ψηφιακή εποχή. Αναφέρεται αυτό στο έγγραφο του Open Up Education και στο σχέδιο κειμένου και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε. Okay. Uh, I I had to go in another. Ναι, ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να παραστώ σε κάποια άλλη επιτροπή και νομίζω ότι έχω φτάσει και στο τέλος, διότι δεν βλέπω άλλους συναδέλφους εδώ να θέλουν να ζητήσουν το λόγο. Ο κύριος Κούρια. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση πολύ σύντομη στους εμπειρογνωμονές μας. Επειδή σχεδόν όλοι επεσήμαναν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, αλλά φαντάζομαι και μεταξύ άλλων χωρών. Θα ήθελα να μου πείτε τι κατά την άποψή σας είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει καταρχάς για να μειώσουμε αυτό το χάσμα δεδομένου ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό είναι δευτερεύον. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των χωρών μας, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όπου υπάρχει διαφορετική νομοθεσία, διαφορετικό επίπεδο ποιότητας της εκπαίδευσης, ε, τόσο για τα σχολεία όσο και για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μπορεί σε κάποιο βαθμό ε, σε σύγκριση με τις Ηνωμένε χώρε του Δητικού Κόσμου να είναι ή με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου να είναι εις βάρος μας. Ε, ποια είναι κατά την άποψή σας τα βασικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ κάτι παρόμοιο θέλω να ρωτήσω, κυρίως για τα σχολεία γιατί στα πανεπιστήμια οι καθηγητές είναι ελεύθεροι σχετικά με το πώς θα διδάξουν, ενώ στα σχολεία είναι πιο περιοριστικά τα πράγματα, πιο ελεγχόμενα. Έχουμε αυστηρά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, διδασκαλίας. Στη Γερμανία Έχουμε βέβαια, στην Ευρώπη έχουμε 28 ε, εκπαιδευτικά ε, ιδρύματα, ε, συστήματα συγγνώμη, και στη Γερμανία κάθε ομόσπονδο κρατήδιο βέβαια έχει τη δική του πολιτική παιδείας με διαφορετικά αποκλήσεις στα περιεχόμενα. Ο κύριος Μέλχερ είπε ότι και η εκδοτική και των σχολικών βιβλίων εκείνοι που ετοιμάζουν ε, με μορφή βιβλίου τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα ε, δεν ε, έχουν εξυγχρονιστεί. Εμείς χρειαζόμαστε και μια πιστοποίηση των καινούριων προγραμμάτων ούτως ώστε να ενταχθούν στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Και πώς μπορούμε με τις ε, δυνατότητες που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή μπορούμε μόνο συντονιστικά να δράσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς με τις αρμοδιότητες που διαθέτουμε, τόσο ώστε να υπάρξει καμιά, κάποια πρόοδος, γιατί στα βιβλία ας πούμε, ε, παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να ε, κυκλοφορήσουν καινούρια βιβλία. Αυτά που έχουμε σε μεγάλο βαθμό είναι απαρχαιωμένα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο. Θα, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι αν είχαμε ψηφιακό περιεχόμενο. Πολύ πιο ευέλικτοι από ό,τι μας επιτρέπουν τα τωρινά βιβλία. Επίσης και σε επίπεδο πιστοποίησης πρέπει να κινηθούμε, ούτως ώστε και οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι στα σχολεία να ξέρουν τι πρέπει να διδάξουν και πώς θα πιστοποιηθεί αυτό. Εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες, αλλά έστω με αυτές πώς μπορούμε να δράσουμε πιο υποστηρικτικά, κυρίως ε, για τα σχολεία και να προωθήσουμε την πρόοδο εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Χαίρομαι που το συζητάμε το ζήτημα αυτό. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, το συζητάμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Αναφερθήκαμε στις διάφορες δυνατότητες ε, για να υπάρχουν ε, ανοιχτά μαθήματα, ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη, ουσιαστικά να ανοίξει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Εάν όμως το θέμα αυτό τεθεί στις προτεραιότητες του θεματολογίου μας, ε, ε, καταφέρνουμε να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προς τα μπρος. Έτσι δεν θα βρεθούμε στα μετόπιστεν ε, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πολύ καλύτερες πλέον οι προϋποθέσεις για να μπορούμε να έχουμε διαλειτουργικότητα, κατάλληλη σύνδεση και εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα χάνει το μονοπολίο του στον τομέα αυτό και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ρηξικέλευτες αλλαγές, νέες ε, διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, οι οποίες θα προκύψουν από την όλη διαδικασία και δεν υπάρχει πλέον ε, ο κεντρικός ρόλος του διδάσκοντος. Παλιά αυτό ήταν το ίδιο το πανεπιστήμιο. Αλλά πλέον οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βρουν πόρους, ε, μπορούν να βρουν τρόπο να διδαχθούν παντού, έξω από το σχολικό χώρο. Ε, η πληροφορική και η τεχνολογία, ε, όλες αυτές οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον κλάδο εκβάθρων. Και οι νέες γενναίες η γενιά του Nintendo μεγαλώνει σιγά σιγά και αυτοί είναι οι αυτόχθονες αν θέλετε, οι πρώτοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την ψηφιακή εποχή. Βεβαίως όταν θα διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους ε, θα αντιμετωπίσουν ίσως κάποιες δυσκολίες διότι λαμβάνουν πληροφορίες από πάρα πολλές πηγές. Ε, αναφέρεται πολλές φορές αυτή η ταυτότητα patchwork, ε, όπου είναι τα πάντα εμβαλωματικά και η, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη πηγή γνώσης. Ε, και φυσικά είναι πολύ διαφορετικές αυτές οι γενιές από τις γενιές που ε, μεγάλωσαν πριν από 30-40 χρόνια, διότι θα πρέπει να λάβουν πάρα πολλές πληροφορίες προκειμένου να μπορέσουν να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους. Έχω και κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με ένα άλλο ζήτημα. Είμαι βέβαιος ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση θα αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό τμήμα των πανεπιστημιακών σπουδών στο μέλλον. Αναφερόμαστε στην τρίτη πλέον γενεά πανεπιστημίων. Πανεπιστήμια τα οποία θα προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα και θα μπορούν να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά θα είναι αυτά τα οποία θα αποφασίζουν πώς θα διαμορφώνεται το μέλλον της παιδείας. Αλλά υπάρχει και το αιώνιο ερώτημα. Χρηματοδότηση και νομικά δικαιώματα. Πώς θα μπορούν τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν κατάλληλα κονδύλια για να αναπτυχθούν αυτά τα προγράμματα και πώς θα επιληθεί το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και των λοιπών δικαιωμάτων. Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα όταν ε, γίνεται συζήτηση για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Einigen Sie sich, wer von Ihnen reden möchte, ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Να πω κάτι για την ερώτηση Ηρίας ε, Καμερέβερτ που ρώτησε για την πιστοποίηση και την επικύρωση των σχολικών περιεχομένων όταν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ψηφιακά μέσα, όχι μόνο στη Γερμανία, γενικά. Αυτό το θέμα εδώ και δέκα χρόνια συζητείται από τους ε, εμπειρογνώμονες των Υπουργείων και των εκδοτικών οίκων. Ακόμη δεν έχει βρεθεί η πιστική λύση που να τη γνωρίζω εγώ τουλάχιστον και θα πρότεινα ε, σε σχέση με αυτό που ρωτάτε το, ότι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα σπρώξει μπροστά αυτά τα πράγματα, να βοηθήσει, να ε, βελτιώσει την νομοθεσία. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ε, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα γνωρίζει την κατάσταση στα κράτη-μέλη και θα καταλήξουν σε μια καινούρια λύση μέσα από ανταλλαγή απόψεων παρακολουθώντας τι γίνεται στα επιμέρους κράτη-μέλη. Υπάρχει μια διαδικασία, ένα μοντέλο που εγώ θα το συνιστούσα επειδή είναι ρευστά τα ψηφιακά περιεχόμενα, επειδή μπορούν να συνδυάζονται πολύ εύκολα και σε μεγάλο βαθμό, και στα πλαίσια των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων που θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ σωστά, με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις δεν θα μπορεί κάθε εκπαιδευτική ενότητα να εγκρίνεται και να πιστοποιείται. Αποκλείεται αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς πια. Άρα λοιπόν θα πρότεινα, και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος που το λέω αυτό, ε, ότι θα πρέπει να πιστοποιούνται επαγγελματίες φορείς που προσφέρουν τέτοια περιεχόμενα που θα αναπτύξουν διαδικασίες ε, για το πώς τα περιεχόμενα που διαθέτουν για τα σχολεία είτε είναι δωρεάν είτε είναι επαμοιβή, αυτά πώς θα πιστοποιούνται ως προς την ποιότητά τους από πριν. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει σε κρατικό επίπεδο. Γίνεται και σε άλλους τομείς άλλωστε. Αντίστοιχο σύστημα διαπίστευσης, για παράδειγμα, έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πολλοί φορείς στον τομέα της επιμόρφωσης πιστοποιούνται με, από αρμόδιες αρχές, από φορείς που καμιά φορά είναι και ιδιωτικοί, αλλά υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο παρόλα αυτά. Έτσι γίνεται η πιστοποίηση και μετά μπορούν να προσφέρουν περιεχόμενα. Το ίδιο μπορεί, και κάτι ανάλογο τέλο πάντων, μπορεί να ισχύσει και για τα ψηφιακά μέσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάλκενμπουργκ θέλει να πει τίποτε. Ορίστε. Ε, thank you. Σας ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση ήταν ε, για την υστέρηση που έχουμε σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το χάσμα. Υπάρχουν αρκετά σημεία εδώ. Καταρχάς, να πω ότι το εκπαιδευτικό μας ε, σύστημα είναι ακόμα πολύ προνομιακό, πολύ καλά οργανωμένο και υπάρχει πολύ καλή χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια. Ακόμα λοιπόν, για πολλά πανεπιστήμια δεν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή έχουν αυτή την πολυτέλεια, γεγονός όμως το οποίο καταδεικνύει και ότι δεν αντιλαμβάνονται ακόμα καλά τι ακριβώς θα συμβεί. Νομίζω ότι με την ε, πρωτοβουλία ε, που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άνοιγμα της ε, εκπαίδευσης έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και έτσι θα μπορέσουν ίσως και πολλά πανεπιστήμια να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, επενδύονται και πάρα πολλά κονδύλια όμως στο θέμα αυτό. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, αλλά και τα πανεπιστήμια αυτά τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν αυτή την οδό. Τα Αμερικανικά πανεπιστήμια επενδύουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια για ε, τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος και μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση προγράμματος εδώ με 300.000 ε, ευρώ. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά και δεν μπορείς να, γίνεις, ε, να γίνει τεράστια αλλαγή με μερικές χιλιάδες ευρώ. Ε, χρειαζόμαστε κάποια μεγαλύτερα προγράμματα που πραγματικά θα αλλάξουν την κατάσταση. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι οι γλώσσες. Για το δικό μου το πανεπιστήμιο δεν υπάρχει πρόβλημα διότι έχουμε επιλέξει ε, ως βασική γλώσσα εργασίας στην αγγλική γλώσσα, αλλά πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν έχουν επιλέξει αυτή την οδό και αυτό φυσικά σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η πρόσβαση ε, και ε, απευθύνονται σε μικρότερο αριθμό φοιτητών. Να σας δώσω και κάποια καλά παραδείγματα Υπάρχει η Open Course Library, η βιβλιοθήκη ε, η οποία είναι πρωτοβουλία της Βοστόνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποφασίστηκε ότι ε, τα χρήματα τα οποία δίνονται για τα βιβλία των φοιτητών θα μπορούσαν ίσως να διατεθούν για να προσφέρονται ανοιχτά μαθήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα πανεπιστήμια ώστε να μπορέσουν να τα προσαρμόσουν στο δικό τους το σύστημα. Και αντί ε, για διδακτικά βιβλία δίνονται πλέον κονδύλια για αυτά τα ανοιχτά μαθήματα. Η πολιτεία έτσι δαπανά λιγότερα χρήματα, οι φοιτητές έχουν πολύ περισσότερη ε, και πιο εύκολη πρόσβαση και σε μαθήματα ε, και ε, πλέον πολλές άλλες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιγράφουν αυτό το σύστημα και ίσως αυτό θα ήταν ενδιαφέρον μοντέλο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης υπήρχε και μια ερώτηση για την απώλεια του μονοπωλίου των πανεπιστημίων. Είπατε ότι περνάμε σε πανεπιστήμια τρίτης γενεάς ε, και υπάρχει θέμα κονδυλίων και νομικών δικαιωμάτων και πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, προσωπικώς θεωρώ ότι πολλά πανεπιστήμια θεωρούν ότι αυτά είναι η αιτία γιατί δεν μπορούν να επιτύχουν τι μπορούν να κάνουν. Ε, εμείς στο Πανεπιστήμιο όμως σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε με το πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε σίγουρα να υπάρχουν πολύ λιγότεροι περιορισμοί, αλλά έχουμε ακόμα πολλές δυνατότητες εντός του παρόντος πλαισίου. Σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων έχουμε ήδη αρκετό περιθώριο να γίνουν αρκετά πράγματα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αν κάποιο αποφασίσει να επενδύσει σε κάτι ω πανεπιστήμιο, πάντα θα βρεθούν κάπου κονδύλια. Υπάρχουν κάποια νομικά προσκόμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ένας φοιτητής θα πρέπει να εδρεύει στη χώρα στην οποία φυτά για να μπορεί να, χρημα... λαμβάνει υποτροφίες για παράδειγμα και θα πρέπει να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Ε, το Υπουργείο Παιδείας στις κάτω χώρες εξετάζει πώς μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας. Ε, φέτος, ε, ε, επειδή είμαστε και πρωτοπόροι, προσπαθεί να δει μαζί μας πώς μπορούμε να τους δώσουμε και περιθώριο να καινοτομήσουμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει κάτι αντίστοιχο. Yes. <clears throat> I try to answer to the whole of the question since there are some First of all, Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να αμφισβητήσω το ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει. Ίσως να ισχύει αυτό σαν μέσο όρο, αλλά βασικά στην Ευρώπη είμαστε σε παίζουμε ηγετικό ρόλο στα MOOCs, τουλάχιστον για τους φοιτητέ που τα παρακολουθούν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, αλλά δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού για τα MOOCs. Υπάρχουν μερικές χώρες που είναι ηγέτιδες επίσης στη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για την παιδεία στην Ευρώπη. Δεν ισχύουν τα ίδια παντού βέβαια. Τρίτον, υπάρχουν προγράμματα ήδη όπως η διδημοποίηση σχολείων από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας αλλά επίσης το GoLab, το Open Discovery Space και άλλα είναι τεράστια προγράμματα με σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για την εκπαίδευση ιδίως θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Είναι προγράμματα που υπάρχουν μόνο στην Ευρώπη και τα ζηλεύουν όλοι. Τώρα, πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι τα τωρινά νομοθετήματα που ισχύουν και που ενέκριναν η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είναι και αυτά ένα τεράστιο βήμα. Πώς θα καταλήξουμε όμως σε αυτά αποτελέσματα. Το κανονικότερο θα ήταν να πούμε πρέπει οι χώρες μέλη που έχουν διαφορές μεταξύ τους να έρθουν όλες στο ίσο, σε ίσο σημείο. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτή η προσέγγιση top-down αλλά και η αντίθετη bottom-up από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους δηλαδή και τα δίκτυα που συμμετέχουν στην εφαρμογή αυτών των νομοθετημάτων στις χώρες μέλη. Υπάρχουν οργανώσεις χριστών, φοιτητών, γονέων κλπ. Διδασκάλων βέβαια. Και όλα αυτά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να πείσουν, για να προωθήσουν, για να διαδώσουν τα αποτελέσματα της, ε, του είδους αυτού της παιδείας. Και έχουμε σχεδόν αγνοήσει τα τελευταία 20 χρόνια έρευνα στον τομέα αυτών. Όταν λέμε δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, έχουμε αλλά μικρότερων αριθμών φοιτητών και προγραμμάτων για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη ενδιαφερόμενοι και φυσικά τα πανεπιστήμια, τα ίδια τα μορφωτικά ιδρύματα. Τα σχολεία ε, ελέγχονται πολύ. Ναι, αυτό συνήθως γίνεται, αλλά έτσι είναι με τα σχολεία, έτσι γίνεται. Πώς θα λειτουργήσουν αλλιώς. Δεν πρέπει να αλλάξουμε όμως το θέμα της ποιότητας. Η ποιότητα μπορεί να υπάρξει και από τον έλεγχο, μπορεί και αλλιώς όμως. Άρα υπάρχει χώρος για μεγαλύτερο άνοιγμα των προγραμμάτων και των συστημάτων όλα όσα ελέγχουμε δεν είναι απαλήτως απαραίτητο να τα ελέγχουμε τέλος. Το κόστος της καινοτομίας. Δεν θα ήταν σωστό βέβαια να πούμε ότι η χρήση της τεχνολογίας για παιδεία είναι ένας τρόπος μείωσης ε, από το δημόσιο τομέα των επενδύσεων στην παιδεία. Ισχύει όμως ότι μια νέα οικονομία της παιδείας μπορεί να φανταστεί κανείς με ειδίκευση και απλοποίηση και αυτό δεν σημαίνει λιγότερους καθηγητές αλλά σίγουρα σημαίνει διαφορετικό ρόλο, διαφορετική οργάνωση, διαφορετικές μορφές συνεργασίας των ε, Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης ώστε να πάψουν πια μερικά να διδάσκουν μόνο τοπικά και άλλα τα πιο γνωστά να είναι μόνο εκείνα που διδάσκουν και ευρύτερα αν επικεντρωθούμε στο θέμα του ότι και τοπικά πανεπιστήμια ε, μπορεί να είναι ε, πολύ σημαντικά. Δεν αρκεί αυτό. Υπάρχουν κέντρα αριστείας, αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν χιλιάδες κέντρα αριστείας. Πρέπει σε μερικά να γίνει κάποια απλοποίηση και εκλογήκευση. Μέσω της συνεργασίας, όχι μέσω καταργήσεων, δεν συστήνουμε αυτό. Λέμε να σκεφτούμε νέους τρόπους συνεργασίας και βέβαια αυτό που θα βοηθούσε την Ευρώπη να προχωρήσει θα ήταν να το προσέξουν το θέμα αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερο να διαδοθεί το νέο αυτό για τα μουξ ας πούμε. Γίνεται συζήτηση για την κινητικότητα των φοιτητών, το έρασμος δηλαδή, αλλά δεν γίνεται αρκετή συζήτηση για άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Ευρώπη, όπως τα MOOCs που βασίζονται στην τεχνολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Περέιρα, ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πω δύο λόγια και μετά ο Μάρκο Μαρσάλα από την DG Connect θα προσθέσει και κάτι ακόμη. Νομίζω ότι η συζήτηση δείχνει σήμερα και αυτό είναι πολύ θετικό σε σχέση με αυτά που κάναμε και εμείς. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες αντιδράσεις σχετικά με το αντικείμενο της συζήτησης. Ε, τώρα το θέμα είναι το πώς θα καταπιαστούμε με το θέμα. Πριν από δύο χρόνια, πριν από ενάμιση χρόνο, ε, είχαμε πολλές συζητήσει ε, που αμφισβητούσαν τη σημασία του θέματος για την Ευρώπη. Οπότε το τελευταίο, το τελευταίο 18 μήνο κάναμε πρόοδο. Έτσι λοιπόν προωθήσαμε τη συζήτηση και παίξαμε και ηγετικό ρόλο. Τώρα, δύο στοιχεία της δράσης μας. Το πρώτο είναι να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε την προσοχή των εμπλεκομένων και των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και υπό αυτή την έννοια, αν και καταλαβαίνουμε ότι όταν η Κομισιόν καταρτήσει συντάξει ανακοίνωση ε, η δυναμική αρχίζει να επιβραδύνεται, όπως είπατε κι εσείς. Όμως παρόλα αυτά η πρόθεσή μας είναι να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτών. Και όπως λέγαμε και συζητούσαμε και με τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια του ανοίγματο της εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, το φθινόπωρο που μας πέρασε, ε, δόθηκε συνέχεια και πολλά θετικά μηνύματα υπάρχουν από την Ιταλική Προεδρία που θα συνεχίσει λέει το θέμα επί Προεδρίας της και θα φροντίσει ώστε και τα κράτη-μέλη να ενταχθούν στις μεταρρυθμίσεις. Για μας η τεχνολογία δεν είναι αυτός σκοπός. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Ντόντι. Θέλουμε καλύτερη πρόσβαση, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ε, αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πνεύμα ε, προχώρησε η Κομισιόν στο άνοιγμα της εκπαίδευσης. Επίσης θέλουμε να με τους εμπλεκόμενους να ευαισθητοποιηθούν για να μιλήσουν περισσότερο και να εστιάσουν περισσότερο στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Ε, δεν μιλώ μόνο για τα κράτη-μέλη εδώ, αλλά πολλούς εμπλεκομένους όπως τους εκδότες. Γιατί αυτό το θέμα των εκδοτών ήταν πολύ σημαντικό στη συζήτηση. Από τότε που αρχίσαμε την πρωτοβουλία, έχουμε ακούσει πολλές οργανώσεις εκδοτών που εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν δύο τρόποι για να δώσουμε συνέχεια σε αυτά που λέγαμε εδώ. Πρώτον, Πρώτος τρόπος, σε σχέση με την ενδεχόμενη επανεξέταση της οδηγίας Infosoc που συζητείται τώρα στους κόλπους της Κομισιόν για να δούμε αν θα ε, προτείνει αναθεώρηση των, ε, της οδηγίας για τα copyrights η Κομισιόν και μέσα στα πλαίσια αυτού του πολύ σύνθετου θέματος και του ευρύτατου θέματος εξετάζουμε και τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού μαθησιακού υλικού και πώς τα copyright επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν την χρήση του ψηφιακού περιεχομένου. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σύνθετη γιατί η shock οδηγία είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι τα θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό και τα ζητήματα δεν θα λυθούν μια νυχτή. Οπότε Φανταζόμαστε ότι αυτή η συζήτηση θα εξακολουθήσει για αρκετούς μήνες ακόμη. Εμείς όμως πάντοτε πιέζομαι για να αναδεικνύουμε τις προκλήσεις του ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού και πώς αυτό συσχετίζεται με το τωρινό πλαίσιο για το copyright. Δεύτερο θέμα που μπορεί να πάρει χρόνο. Συζητήσαμε το τι θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή νομοθεσίας. Συζητήσαμε και με εκδότες και με άλλους ενδιαφερόμενους και εμπλεκομένους για θέματα ε, προτύπων διαλειτουργικότητας για τα περιεχόμενα, επί παραδείγματι, και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πλατφόρμα διευκολυντική για να βρούμε και άλλες λύσεις. μετά την, και, την έγκριση της ανακοίνωσης θα μπορέσουμε πριν από το καλοκαίρι να υποβάλλουμε σε αυτά τα θέματα συγκεκριμένες λύσεις. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω που δεν αφορά μόνο την ε, ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, αν θέλετε, κρατών μελών και άλλων εμπλεκομένων, αλλά και ε, παροχή ε, κινήτρων και μέσα από το έρασμο ΣΥΝ να ε, προωθηθεί η καινοτομία σε αυτό το τομέα. Και εδώ, στα πλαίσια του νέου προγράμματος, θα αναφέρω ε, δύο συγκεκριμένες και πολύ συγκε... Ε, θετικές ευκαιρίες που εγκρίθηκαν και με την συνδρομή του Κοινοβουλίου και αφορούν τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις ή συμπράξεις, στρατηγικές συμπράξεις δηλαδή τομεί που αφορούν την καινοτομία στην εκπαίδευση και τη χρήση τεχνολογιών για αυτήν την καινοτομία υποχρεώνουν ε, την δημιουργία συμπράξεων και τώρα μάλιστα ε, υπάρχει και προκήρυξη διαγωνισμού μέχρι το Μάρτιο και μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι πρωτοβουλίες βάσης θα μπορέσουν να διαμορφωθούν αφού θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος, θα το έχει δημιουργήσει το πρόγραμμά μας. Ε, στο πρόγραμμα υπάρχει μια διεθνής διάσταση, δεν ε, ε, περιοριζόμεθα σε περιφέρειες, θέλουμε συμπράξεις διασυνοριακές και δεύτερον αυτές οι συμπράξεις θα πρέπει να ε, έχουν θετικό αντίκτυπο. Μια επίπτωση θετική, στρατηγική επίπτωση χρειαζόμαστε ε, σχετικά με το πώς εφαρμόζονται ε, τα αποτελέσματά μας στα σχολεία, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις για να υποστηριχθούν οι προτάσεις. Αλλά έτσι μπορούμε να διευρύνουμε την υποστήριξή μας, δηλαδή να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μέσα από τη χρήση τεχνολογίας, να αναζητηθούν εταίρικες και συμπράξεις μέσα το καλύτερο περιεχόμενο ή κάποια πανεπιστήμια που θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας τους, το επιχειρησιακό μοντέλο. Πολλοί τομείς, ενδιαφέροντες τομείς ανοίγονται εδώ. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε θετική επίπτωση με τα λεφτά που δίνουμε. Τέλος, ε, πολιτι... Ε, πειραματισμοί πολιτικής. Και εδώ προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια σχόλια που έγιναν και εδώ σήμερα σχετικά με την αναβάθμιση των ε, επενδύσεων. Οι πειραματισμοί πολιτικής θα είναι project και αυτά, προγράμματα, στον οποίο, στα οποία επικεφαλής θα είναι εθνικές αρχές που θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε επίπεδο σχολείων ή εκπαιδευτικών ε, ιδρυμάτων, που θεωρούμε ότι είναι αρκετά ευρείας βάσης και η προκήρυξη του διαγωνισμού που έχουμε εξετάζει ε, κυρίως τις εγκάρσιες δεξιότητες και τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνολογία για να αξιολογήσουμε οριζόντιες δεξιότητες και τεχνολογίες ε, πληροφορίας και επικοινωνίας. Επίσης ένα πλεονέκτημα της νέας δομής του προγράμματος είναι ότι υπάρχει μεγάλη ευελιξία σε αυτό και θα δείτε ότι και στο πρόγραμμα εργασίας του 2014 αλλά και στις ε, προκηρύξησε για τη χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση για πιο ε, καινοτόμα παιδαγωγικά προγράμματα. Όλες αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν, έχουν έντονη παρουσία σε σχέση με το τι ίσχυε στα παλιά εκπαιδευτικά προγράμματα και τα παλιά μαθησιακά προγράμματα. Τέλος, τρία θέματα που αναφέρατε κι εσείς εδώ, γιατί ε, κάποιος ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, σε τομείς που είμαστε καλοί και μπορούμε να είμαστε στο προσκήνιο. Έχουμε μια ε, ιστορία, μια παράδοση ε, στην αμοιβαία αναγνώριση και τη διαφάνεια των ε, προσόντων και των δεξιοτήτων. είναι δύσκολη διαδικασία η διαδικασία της Μπολόνια υπάρχει εδώ και κάποιες δεκαετίες και παρόλα αυτά δεν έχουν εξαλειφθεί οι δυσκολίες. Είναι εδώ, έχουμε όμως εδώ έναν τομέα όπου η Ευρώπη είναι πιο εξελιγμένη από τι άλλες περιοχές του κόσμου και θα ήταν ενδιαφέρον να αξιοποιήσουμε την πείρα που έχουμε για να δούμε πώς η ψηφιακή μάθηση ή η επιγραμμική όπως λέμε online μάθηση μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτές τις διαδικασίες το θέμα της αναγνώρισης ε, των δεξιοτήτων που ε, επιτυγχάνονται και κατακτώνται επιγραμμικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες διαφάνειας και αναγνώρισης που ήδη διαθέτουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει, που άλλες περιοχές στον κόσμο δεν το έχουν κατακτήσει. Ε, ένα δεύτερο στοιχείο αφορά το ζήτημα της πιστοποίησης των ΑΕΠ και η διαπίστευση για επαγγελματίες φορείς που παρέχουν αυτά τα, τους σπόρους. Εκεί οι απόψεις των διεμπειρογνώμων μας ήταν λίγο διαφορετικές, γιατί είπαμε ότι πρέπει να υπάρχουν οι επαγγελματίες που να διαπιστεύονται, να προβλέπεται διαπίστευσή τους. Ε, μετά είπαμε ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε τα πάντα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρώπη, δηλαδή αυτό που πιστεύουμε, είναι ότι μπορούμε να προσθέσουμε παραμέτρους ποιοτικέ χωρίς να θέλουμε να τις επιβάλλουμε όμως, να υπάρχει δηλαδή μια, ένας κοινό παρονομαστή σχετικά με το τι είναι η ΑΕΠ ποιότητα, χωρίς να περιορίζουμε την παραγωγή των ΑΕΠ, γιατί αυτή είναι η ομορφιά των ΑΕΠ. Είναι ότι είναι αυθόρμητη η παραγωγή τους, είναι από κάτω προς τα πάνω, δεν είναι ελεγχόμενη και ε, προδιαγεγραμμένοι και οι ΑΕΠ μπορούν να εμφανίζονται αντικατοπτρίζοντας τις τάσεις της κοινωνίας. Οπότε από αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι κάποια ποιοτικά πλαίσια μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς όμως να επιβάλλουν και να υπαγορεύουν συστήματα διαπίστευσης ή αυστηρά πλαίσια. Τέλος, κάτι που νομίζουμε ότι ακόμα εκρεμεί και ακόμα το παρακολουθούμε είναι το θέμα των επιχειρησιακών μοντέλων, business models. Το είπατε και εσείς ότι, αν σας κατάλαβα καλά, στην Ολλανδία ένας ε, φοιτητής ε, μπορεί να υποστηρίζεται αν παρακολουθεί ένα μάθημα στην Ολλανδία. Τώρα, με τα επιγραμμικά λεγόμενα online, τα γεωγραφικά όρια καταργούνται. Οπότε πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός θα εξακολουθεί να τα καλύπτει τα μαθήματα αυτά. Αυτά τα θέματα ακόμα είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά για κάποιους μήνους, μήνες ακόμη. Εμείς θα συνεχίζουμε να τα μελετούμε μαζί με τους υπουργούς γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος όπου θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση της μάθησης που γίνεται διαδικτυακά. Και κάποιος ζήτησε και κάποια στοιχεία αριθμητικά. Στα MOOCs αυτά τα μαζικά διαδικτυακά μαθήματα κάποιοι είπαν ότι είναι μια μόδα που θα εξαφανιστεί. Ε, συμφωνούμε με τους προηγούμενους μιλητές ότι ήρθαν για να μείνουν αυτά τα MOOCs γιατί τώρα ε, μαζικοποιείται η τεχνολογία και επιτρέπει να μονιμοποιηθούν κάποια τέτοια φαινόμενα αλλά ε, βέβαια μπαίνουν και ζητήματα πιστοποίησης όπως σας είπα και πριν. Τώρα, κάποια νούμερα που έχει η Κομισιόν. Σήμερα έχουμε 1.369 μουξ. Από αυτά 394 είναι ευρωπαϊκά. Δηλαδή το 1 τέταρτο περίπου, λίγο πάνω από 1 τέταρτο είναι ευρωπαϊκά. Αυτό δείχνει ότι από την πλευρά της προσφοράς δεν είμαστε ε, πρωτοπόροι, μπορεί να είμαστε στην πλευρά της ζήτησης, ότι οι Ευρωπαίοι δηλαδή είναι μεταξύ των μεγαλύτερων χρηστών των ΜΟΚΣ. Κάνουν χρήση αυτών των μαζικών διαδικτυακών ανοιχτών μαθημάτων. Οπότε υπάρχει ανάγκη η Ευρώπη να μάθει περισσότερα για τις εξελίξεις. Όχι μέσα από μια αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, μπορεί να μην χρειάζεται να πάντοτε να πληρώνει για όλα αυτά. Όταν υπάρχει ζήτηση υπάρχει λόγος για να τα συζητάμε όλα αυτά. Και σίγουρα η τάση αυτή δεν θα σταματήσει. Και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τα σχόλια και την ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Και για να συμπληρώσω αυτά που είπε η συνάδελφος, είναι πολύ σημαντικό να γίνει καλύτερη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχουμε συγκεντρώσει τα τελευταία 20 χρόνια. Αναγνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει συνεχής καινοτομία και έρευνα και το νέο πρόγραμμα πλαίσιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει ε, σε θέματα έρευνας και καινοτομίας αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, καθώς και τα πιο μεγάλη κλίμακας προγράμματα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της γνώσης, διάχυση της γνώσης, ώστε να μπορέσει αυτό να συνεισφέρει ε, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτές τις ε, ρηξικέλευτες ε, ε, εξελίξεις που έχουμε στην τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν άκουσα αυτά που είπατε στην αρχή, αλλά η συζήτηση έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταπιάστηκε με ένα θέμα το οποίο φαίνεται πολύ δύσκολο να το ε, πραγματοποιήσει. Ε, στην αρχή το βουνό μας φαίνεται πολύ δύσκολο να το ε, να, να αναρριχηθούμε, αλλά μετά τα καταφέρνουμε. Υπάρχουν έτσι μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται τώρα, ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν αξιοποιήσιμες. Αυτό το αναξιοποίητο δυναμικό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε παντού, να το εκμεταλλευτούμε παντού. Και στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις επαγγελματικές σχολές, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πάνω απ' όλα. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω το είπατε αρκετές φορές και εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να το συζητήσουμε να το προωθήσουμε, να το δημοσιοποιήσουμε, να κερδίσουμε το ενδιαφέρον άλλων, οι εμπλεκόμενοι, οι stakeholders που είναι και δικτυωμένοι, που τους αναφέρατε, θα φροντίσουν ο καθένας στη χώρα του, ούτω ώστε να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες και οι δυνατότητες που υπάρχουν και να ε, συναγάγουν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές ελπίδες που συνδέονται εδώ σε αυτό το τομέα. Πολλά πρέπει να γίνουν. Βέβαια δεν θα κινηθούμε μόνοι μας, ε, δεν θα, καταφέρουμε, θα τα κάνουμε εμείς αυτά. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή να ε, ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό. Είμαστε περιορισμένοι και από τη συνθήκη της Λισαβόνας και όπως και του Μάστριχ. Επικουρικά μόνο εδώ ε, δραστηριοποιούμεθα. Αλλά θα ήταν ανόητο αν δεν λαμβάναμε υπόψη μας τις γνώσεις της τεχνολογίας, τα, τα καινούργια δεδομένα. Είναι, θα ήταν ανόητο να μην τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία σε όλους τους τομείς. Εύχομαι να πάει καλά, να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό και να συμφωνήσει και το Συμβούλιο των Υπουργών, ώστε να τεθεί στην ημερήσια διάταξη και με τους Υπουργούς Έρευνας ε, ο καθένα στη χώρα, το κάθε υπουργό παιδεία πρέπει να το ε, συζητήσει το θέμα. Δεν τελειώνει η υπόθεση αυτή με αυτή την ανακοίνωση. Ή τώρα αρχίζει ε, και θα κρατήσει πολύ. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι θα κάνουμε μεγάλα βήματα άμεσα. Καλό είναι να κάνουμε και μικρά βήματα. Καλά είναι και αυτά και να λάβουμε υπόψη μας και ορισμένα θέματα όπως αυτά που είπατε, δηλαδή δικαιώματα δημιουργού κλπ, ε, πνευματική ιδιοκτησία κλπ. Ε, στη Γερμανία, για παράδειγμα, στον τομέα των βιβλιοπολίων, δηλαδή εμπόριο βιβλίων, εκεί θα υπάρξει κατακραυγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα η οποία τώρα χάνεται. Υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχουν ε, πολλά που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιοριστούμε στα τεχνικά τεχνολογικά θέματα. Είναι λίγο και ολισθηρό το ε, πεδίο. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, ευχαριστώ για την παρουσία σας σε αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που έδωσε αυτή τη γερή σπροξιά και εύχομαι να έχουμε καλή επιτυχία. Φτάσαμε στο τέλος της ακρόασης. Και μου φαίνεται φτάσαμε και στο τέλος της συνεδρίασης. Μάλιστα. Μετά θα συνεδριάσουμε οι συντονιστές. Αύριο.